Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε σας παρακαλώ για να αρχίσουμε αμέσως τη συνεδρίασή μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε θερμά στο δεύτερο τμήμα της σημερινής μας συνεδρίασης της Επιτροπής Γεωργίας. Ευθύς εξ αρχής θα ήθελα να ε, περάσουμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Γεωργίας ε, και Δασών, προεδρεύοντα του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας, τον ε, Υπουργό τον κύριο Λέπα. Καλωσορίσατε θερμά, κύριε Προεδρεύον, κύριε Υπουργέ, στην Επιτροπή μας. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε ε, ως Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ακούσουμε τις προτεραιότητες της Φιλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου στον τομέα της Γεωργίας ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής για τη χρηματοδότηση ε, της δημοσιονομικές προοπτικές. Και φυσικά ενδιαφερόμαστε και για τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, παράδειγμα Mercosur και άλλες. Νομίζω ότι ε, είναι αυτά τα θέματα που συγκεντρώνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προτεραιότητα ε, αποτελούν στην Επιτροπή μας. Ε, θα σας δώσω αμέσως το λόγο για να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητες της Προεδρίας και στη συνέχεια θα πάρουν το λόγο οι ε, συντονιστές σε ένα πρώτο γύρο, τα γνωρίζουν αυτά οι συνάδελφοι. Θα ακολουθήσει ένας πρώτος γύρος απαντήσεων και στη συνέχεια οι υπόλοιποι συνάδελφοι, τα μέλη της Επιτροπής. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Ως ε, υπουργό Αρμόδιος για τη Γεωργία και τα Δάση, χαίρομαι ιδιαίτερος ε, που έρχομαι στην Επιτροπή σας για να σας μιλήσω για τους στόχους και τις προτεραιότητες της Φιλανδικής Προεδρίας και πώς σκοπεύουμε να το υλοποιήσουμε. Ο διάλογος μεταξύ των κοινοτικών θεσμικών οργάνων έχει μεγάλη σημασία και σημερινή συνάντηση είναι εξαιρετικό παράδειγμα και χαρακτηριστικό του επικοδομητικού διαλόγου που θέλουμε να προωθήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας. Εσείς είστε ε, αίρετοι άμεσα εκλεγμένοι από τους Ευρωπαίους πολίτες και φυσικά προσπίζετε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και τις κοινέ ε, ευρωπαϊκές μας αξίες. Το έργο σας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είχαμε ε, θαυμάσια εμπειρία αγαστή συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη Φιλανδία και αυτό περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη σημερινή συζήτηση και τις ερωτήσεις που θα θέσετε. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας εκφράσω κάποιες σκέψεις μου για τις προτεραιότητες της Φιλανδικής Προεδρίας. θα επικεντρωθώ σε θέματα που ενδιαφέρουν κυρίως στην Επιτροπή σας. Η Φιλανδική Προεδρία συμπίπτει με ένα σημείο καμπής θεσμικό. Την αλλαγή τη κοινοβουλευτική την αλλαγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την αλλαγή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι διαπραγματεύσει του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, το Brexit, θα δημιουργήσουν νέε προκλήσει και πολύ σοβαρές προκλήσεις ε, και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Στη διάρκεια της Προεδρίας μας θέλουμε να προωθήσουμε την καταπολέμηση, την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, το κράτος δικαίου και τις κοινέ μας ευρωπαϊκές αξίες. Επίσης θέλουμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα σε μια κοινωνικά συνεκτική Ευρώπη. Η Προεδρία μας θα καθοδηγηθεί από την αρχή του ανοίγματο τη εμπιστοσύνη, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα και αηφορία. Η Φιλανδία θα είναι η πρώτη Προεδρία που θα εφαρμόσει έμπρακτα το νέο στρατηγικό πρόγραμμα του Συμβουλίου που στη, τον Ιούνιο. Και φαίνεται και στα, στα προγράμματα των ε, επίσημων και άτυπων ε, Υπουργικών Συμβουλίων. Έχουμε πολύ σημαντικά θέματα επιτάπητος για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλούμαστε να δώσουμε απαντήσεις ε, σε πολλά. Και σίγουρα οι συζητήσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα έχουν μεγάλη σημασία και θα επηρεάσουν την πρόοδο στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Θα πρέπει να βρούμε μια σταθμισμένη, ισορροπημένη απόφαση για το ΠΔΕΛΤΑΠΗ που θα λαμβάνει υπόψη τις παραδοσιακές πολιτικές και τις νέες προκλήσεις. Αυτό θα είναι από τα βασικά μας μελήματα. Επίσης, για να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές θα πρέπει να λάβουμε πολύ σημαντικά μέτρα και να συμφωνήσουμε στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές μας γι' αυτό κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Θα πρέπει επίσης να δούμε πώς θα καταφέρουμε μέχρι το 2050 να υλοποιήσουμε το στόχο μας για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Μάλιστα θα έχουμε στα τέλη του μήνα ένα άτυπο Συμβουλίο Γεωργίας στο Ελσίνκι για τη δέσμευση και αποθήκευση του, φάρο, του άνθρακα στη Γεωργία. Η δέσμευση άνθρακα είναι από τα βασικά μέτρα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα και να αξιοποιηθεί για να μειωθούν οι εκπομπές άνθρακα από τη Γεωργία. Και γι' αυτό θα θέσουμε το ζήτημα στο άτυπο Συμβούλιο Γεωργίας που θα λάβει χώρα στο Ελσίνκι. Επίσης θέλουμε να προωθήσουμε τις συζητήσεις ε, και να ενθαρρύνουμε τους γεωργούς να λάβουν μέτρα για την ε, αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα από τις γεωργικές δραστηριότητες. Επίσης θα πρέπει να διαφυλάξουμε και την βιοπικιλότητα, κάτι που είναι κοινό μας συμφέρον και των γεωργών και των υπολείπων. Η κοινή γεωργική πολιτική βρίσκεται το επίκεντρο της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Έτσι θα εξασφαλίσουμε το βιοπορισμό των γεωργών, λογικές τιμές καταναλωτή, ισορροπημένες αγορές και επίσης ε, μία ασφάλεια ε, τροφικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο βασικός μας στόχος, η παραγωγή τροφίμων, δεν θα πρέπει που να τεθεί σε κίνδυνο. Επίσης, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κερδοφορία τη Ευρωπαϊκή Γεωργία και να λάβουμε υπόψη και τους διεθνείς κανόνες ανταγωνισμού. Ο στόχος της μεταρρύθμισης τη ΚΑΠ είναι να γίνει πιο βιώσιμη η γεωργία και για τον γεωργό αλλά και για το περιβάλλον. Και η πρόοδο ε, στι συζητήσει για τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ είναι από τι βασικέ προτεραιότητε τη Φιλανδική Προεδρία. Γι' αυτό θα ήθελα να επισέλθω σε πιο διεξοδική ανάλυση των στόχων μα. Θέλουμε να σημειώσουμε όσο περισσότερη πρόοδο γίνεται στι διαπραγματεύσει και, άμα μα το επιτρέψει η κατάσταση, να καταλήξουμε και σε μια γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο για τη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική. Οι προηγούμενε προεδρίε έχουν προλιάνει το έδαφο αρκετά, αλλά θα πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις στο Συμβούλιο, ιδιαίτερα για τη φιλοπεριβαλλοντική αρχιτεκτονική της ΚΑΠ και το νέο μοντέλο ε, παρουσίαση αποτελεσμάτων, το delivery model που λέμε. Θα πρέπει να αναζητήσουμε συμβαστική λύση στη διάρκεια της Προεδρίας μας για τα θέματα αυτά. Θέλουμε η Γεωργία να θεωρηθεί ως τμήμα της λύσης για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και όχι ως πρόβλημα. Και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στη μελλοντική ΚΑΠ. Η αρχή της απλούστευσης επίσης αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και θα πρέπει να γίνει σεβαστή σε όλες τις φάσεις ε, της χάραξης, από τη χάραξη μέχρι την εφαρμογή της ΚΑΠ. Επίσης θα πρέπει να σεβαστούμε τη διαφορετική κατάσταση που ισχύει στα κράτη-μέλη και γι' αυτό με το νέο μοντέλο παρουσίασης αποτελεσμάτων, το delivery model, έχουμε περισσότερες ευκαιρίες για κάτι τέτοιο. Θέλουμε οι γεωργοί να έχουν μια σαφή εικόνα για το μέλλον, να μπορούν να έχουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τις γεωργίες τους. Γι' αυτό και θέλουμε να συμφωνήσουμε για τη μεταβατική περίοδο, για την μεταρρυθμιστικά από το συντομότερο δυνατόν. Και ελπίζω να συμφωνήσουμε με το Κοινοβούλιο για την μεταβατική περίοδο, ώστε οι κανόνες να ισχύσουν ήδη από το 2021 και να ξεκαθαρίσει το τοπίο και για τους γεωργούς και για τα κράτη-μέλη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, η Φιλανδία ήταν ανέκαθεν δραστήρια σε θέματα δασών και δασοπονίας και αυτό ισχύει φυσικά και για τη δική μας Προεδρία. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δάση είναι πολύ σημαντικό εργαλείο και γι' αυτό θέλουμε μια πιο συνεπή και συνεκτική πολιτική που θα επηρεάζει θετικά την κατάσταση των δασών. Βρισκόμαστε σε διαδικασία χάραξη μιας νέας στρατηγικής για τα δάση για την περίοδο μετά το 2020. Θα βάλουμε τα δυνατά μας ώστε η νέα στρατηγική να είναι πιο αποτελεσματική από την προηγούμενη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ήταν ανέκαθεν υπέρ τη στρατηγική των δασών και συνέβαλε στη διαμόρφωσή τη και ελπίζω αυτό να ισχύσει και για τη μελλοντική μας στρατηγική για τα δάση. Η κατάσταση των δασών παγκοσμίω είναι ένα επίκαιρο και πολύ σημαντικό θέμα. Ακούσαμε πολύ ενισχυτικέ ειδήσει για τις δασικές πυρκαγιέ στη Βραζιλία πρόσφατα και γενικώ οι πυρκαγιέ στα δάση έχουν αυξηθεί παγκοσμίω. Στη διάρκεια τη πυρκαγιά στην Αμαζονία έχουμε πολλού παράγοντε που συνέβαλαν. Και μάλιστα η αύξηση της γεωργικής, των γεωργικών εκτάσεων είναι από τους παράγοντες που όξυναν το φαινόμενο των πυρκαγιών. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε και από την Φιλανδική Προεδρία να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ήδη προσφερθήκαμε να βοηθήσουμε τη Βραζιλία να κατασβέσει τις πυρκαγιές. Το σημαντικό όμως και αυτό που προέχει είναι να αποτρέψουμε ε, την συνέχιση της αποψήλωσης των δασών στο, στο μέλλον. Τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια ανακοίνωση για τα δάση και την αποψήλωσή τους και η δημοσίευση αυτή περιέχει βασικούς άξονες για την προστασία των δασών παγκοσμίω. Επίσης, χάρη στην ανακοίνωση αυτή, θα μπορέσουμε να προωθήσουμε κάποιες κοινέ δράσει για να ενισχύσουμε την αηφόρο χρήση και διαχείριση των δαζών και να αποτρέψουμε την αποψήλωση ενισχύοντας την αναδάσωση. Μάλιστα, θα προτείνουμε και συμπεράσματα στο Συμβούλιο στη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας για τη στρατηγική των δασών. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη διάρκεια της Φιλανδική Προεδρίας παρακολουθούμε στενά και το Συμβούλιο τι ε, διεθνεί εμπορικές διαπραγματεύσεις και την κατάσταση στις γεωργικέ αγορέ. Στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλίας του Ιουλίου συζητήσαμε την Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μερκοσούρ η συμφωνία αυτή δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ικανή να προωθήσει ένα ελεγχόμενο σύστημα, διεθνές εμπορικό σύστημα που θα εδράζεται σε κανόνε. Στην παρούσα κατάσταση, μια τέτοια συμφωνία δεν είναι κάτι αυτονόητο. Η οικονομική συμφωνία και η σημασία, τη της ε, εμπορικής αυτής συμφωνίας είναι τεράστια. Μάλιστα, συζητήθηκε εκτενώς ε, και στα κράτη-μέλη και στη δημόσια συζήτηση και επηρεάζει ιδιαίτερα τη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η επίδραση ε, δημιούργησε ανησυχίες. Επίσης, ε, οι πυρκαγιές στη Βραζιλία έγιναν κάποια ερωτήματα ως προς την αποψήλωση του Αμαζονίου και το συσχετισμό τους με τη Συμφωνία Μερκοσούρ. Σίγουρα η κατάσταση ε, των γεωργικών αγορών σε ευαίσθητους τομείς όπως είναι τα πολερικά, το βόλιο και η ζάχαρη θα πρέπει να παρακολουθούνται εκ του σύνεγγης. Πάντως με τη συμφωνία θα ενισχυθεί η συνεργασία και η διαφάνεια και σε θέματα φυτογενομικά. Το ευρωπαϊκό μοντέλο δράσης δεν θα αλλάξει, σας διαβεβαιώ. Και τα εισαγόμενα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο μέλλον θα πρέπει να πληρούν τις υγειονομικές και φυτοϊγειονομικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται να κάνουμε καμία παραχώρηση εδώ. Η Συμφωνία Μερκοσούρ περιλαμβάνει και ένα τμήμα για την αηφόρο ανάπτυξη και τη δέσμευση ε, της εφαρμογής της Συμφωνίας των Παρισίων. Επίσης, ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποψήλωση εφόσον συμφωνηθεί η Συμφωνία εφόσον ε, ε, υλοποιηθεί η συμφωνία και όλα τα συμβαλωμένα μέρη θα πρέπει να την τηρήσουν πιστά. Η Ευρωπαϊκή Γεωργία προτείνει υψηλής, παράγει υψηλή ποιότητα τρόφιμα και μάλιστα με υπεύθυνο τρόπο. Στο μέλλον όμως θα ήθελα περισσότερες δράσεις για να ενισχύσουμε την ε, πρωτεϊνική μας επάρκεια και την επάρκειά μας σε πρωτεΐνοχες καλλιέργειες. Έτσι θα γίνει και η παραγωγή πρωτεϊνών πιο βιώσιμη και αηφόρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, το θέμα της αφρικανικής πανόλης των χείρων θα το παρακολουθήσουμε στενά, γιατί η εξάπλωση της ζωνόσου αυτής στην από και στην Κίνα πήρε μεγάλες διαστάσεις, κάτι που μας προβληματίζει. Ε, και θα το συζητήσουν αυτό επικεφαλή των ιατρικών υπηρεσιών το Σεπτέμβριο στο Ελσίνκι. Ε, μας ενδιαφέρει και η καλή μεταχείριση των ζώων, η ευζοία. Εσείς ε, συμμετείχατε με τα ψηφίσματά σας στην, στον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής και τα δύο θέματα είναι σημαντικά για την προώθηση μιας αηφόρου κτηνοτροφίας. Επίσης, οι μεταφορές ζώων σε μεγάλη απόσταση είναι πολύ σοβαρό θέμα. Όταν έχουμε μεταφορά των ζώων σε μεγάλε αποστάσει και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα με υψηλέ θερμοκρασίε που υπερβαίνουν τα αποδεκτά όρια ε, και σε εμπορευματοκιβώτια, στεγανά κλειστά, μια τέτοια κατάσταση είναι απαράδεκτη από άποψη καλή μεταχείριση των ζώων. Επίση, η μικροβιακή εντοχή είναι μια παγκόσμια απειλή και θα πρέπει να την επιβραδύνουμε. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει δραστήριο ρόλο παγκοσμίω για να σημειωθεί πρόοδο στο θέμα της καταπολέμησης της μικροβιακής αντοχής. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτές ήταν οι βασικές προτεραιότητες της ε, φιλανδική προεδρία στη Γεωργία και τα δάση. Σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μου δώσετε να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση και περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον και αντιμονία τη συζήτηση και τις ερωτήσεις σας σε ό,τι αφορά τους κοινούς μας στόχους, δηλαδή την επίτευξη μιας αηφόρου γεωργίας, αηφόρων δασών, αηφόρου δασοκομείας και τη βελτίωση της κατάστασης των γεωργών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά, Υπουργέ, για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων σας πολλές οι προτεραιότητες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην υλοποίηση όλων αυτών των στόχων που έχετε θέσει το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες. Αρχίζουμε τώρα λοιπόν από τους συντονιστές. Πρώτος είναι ο κύριος Ντόρφμαν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Υπουργέ ε, για την σημερινή σας παρουσία στην Επιτροπή μας για να σας παρουσιάσετε τις προτεραιότητες και τις προτάσεις Προεδρίας οι στόχοι της νέας κοινή γεωργικής πολιτικής μας βρίσκουν σύμφωνο σε μεγάλο βαθμό και κυρίως το θέμα πώς θα απλουστεύσουμε τη γεωργική πολιτική ε, για τους γεωργούς, τους αγρότες, αλλά και για τις διοικήσεις. Αυτό είναι τεράστια πρόκληση. Πιστεύω όμως επίσης ότι στη δική σας προεδρία Υπάρχει επίσης κάτι πολύ σημαντικό που είναι το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο που σας έχει πέσει ο κλήρος. Η πρόταση αυτή τη στιγμή για τη γεωργία κατά την άποψή μου δεν είναι ικανοποιητική. Και για να έχουμε ικανοποιητική πρόταση θα πρέπει να αυξήσουμε συνολικά την βρικοδότηση του PDP. Ιδιαίτερα είναι διαφορετικές ε, οι περικοπές που έχουν γίνει στον πρώτο και στο δεύτερο πυλώνα, οι πολύ μεγαλύτερες στο δεύτερο πυλώνα. Και αυτό το θεωρώ ιδιαίτερα προβληματικό και με ενδιαφέρει ε, να μου πείτε την άποψή σας γιατί η χώρα σας, η Φιλανδία, είναι μια χώρα που παίζει ιδιαίτερο ρόλο ε, ο δεύτερος πυλώνας. γιατί πολλοί γεωργοί έχουν ε, ε, εδάφη και γέες που πρέπει να καλλιεργηθούν υπό πάρα πολύ αντίξωες καιρικέ συνθήκες και άλλες. Και είναι ε, για μένα ε, σημαντική η γνώμη σας. Συμφωνώ για όσα είπατε για τη στρατηγική για τα δάση. Πριν από ένα χρόνο και κάτι είχαμε πάει και στη χώρα σας, στην κεντρική Φιλανδία και είδαμε διάφορες ε, δασοκομικές μονάδες. Μας εντυπωσίασε πάρα πολύ αυτό και πώς μπορεί κανείς να ε, ασκεί μια βιώσιμη δασοκομεία. Η προστασία και η βιωσιμότητα και η εκμετάλλευση των δασών συμβαδίζουν εκεί και μπορεί να γίνει αυτό με τρόπο λογικό και βιώσιμο. Και αφού τέλειωσε και ο χρόνος μου, ένα τελευταίο που δεν ε, αναφερθήκατε σε αυτό, ε, αλλά ε, είναι ίσως τη δική σας αρμοδιότητα έμασα. Είναι τα μεγάλα σαρκοβόρα θηλαστικά, οι αρκούδες και οι λύκοι και περιμένουμε σε λίγες εβδομάδες κάποια αποτελέσματα. Ε, μπορείτε με τον συνάδελφο Υπουργό Περιβάλλοντος να το θέσετε στο Συμβούλιο αυτό για να το προωθήσουμε αποτελεσματικά, γιατί εδώ και χρόνια μας απασχολεί. Γιατί δεν έχει κάνει και τίποτα ο αρμόδιο επίτροπο. Χρειάζεται επιγόντω μία πρόταση στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Ντόρφμαν, αν είναι δυνατόν να τηρείτε το χρόνο, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να φύγει ο Υπουργό, ο κύριος Δικάστρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για την ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε. Θα είμαι σύντομος, θα τηρήσω το δίλεπτο. Είπατε ότι οι μεταρρυθμίσεις που παρουσίασε ο Επίτροπος Χόγκαν ε, σκοπό έχουν να κάνουν πιο βιώσιμη την ΚΑΠ ενισχύοντας τα περιβαλλοντικά μέτρα και διεγείροντας σε μία ενάρετη, θα λέγαμε, συμπεριφορά από τους αγρότες. Συμφωνούμε, αλλά το δεύτερο βήμα είναι να απλουστεύσουμε την εφαρμογή της ΚΑΠ, μειώνοντας τη γραφειοκρατία για τους αγρότες. Η ερώτηση λοιπόν προς εσάς είναι, πιστεύετε ότι έχουν υλοποιηθεί αυτοί οι στόχοι. Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης, πιστεύετε ότι αν τα κράτη-μέλη θα είναι τα μόνα υπεύθυνα για το σχετικά με την απόφαση πότε θα παρέμβουν είναι σωστό από άποψη περιβαλλοντική και απλουστευτική. Δεν νομίζετε ότι πρόκειται για μια επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ ή δεν υπάρχει ο κίνδυνος επανεθνικοποίησης που θα δημιουργήσει με τη σειρά του στρεβλώσεις στη συμπεριφορά. Ε, ε, νομίζω ότι η φάση μετάβασης είναι σημαντική. Την περιμένουμε. Και βέβαια η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να εφαρμοστεί ε, χωρίς αυτή το, την 1η Ιανουαρίου του 2021. Καλό θα ήταν αν κατά την Προεδρία σας λοιπόν ε, τα, το, η πράξη για τη μετάβαση θα μπορούσε να παρουσιαστεί για να υπάρχει και ασφάλεια για τους αγρότες και να έχει και καλή, θετικό αντίκτυπο στην ΚΑΠ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Υπουργέ Λέπα, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Εναποθέτουμε μεγάλες ελπίδες στη Φιλανδική Προεδρία, γιατί γνωρίζομαι ότι εργάζεστε δομημένα και στοχευμένα. Ε, βέβαια, το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι σημαντικό, το Brexit επίσης. Υπάρχουν πολλές ε, άγνωστες παράμετροι, αλλά πολύ σημαντικό θα είναι στη συζητήση μας ε, το θέμα της Γεωργίας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε υπέρ της ε, παραγωγής ε, τροφίμων ε, στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί τους αγρότες που θέλουν βέβαια σχεδιασμό, απλούστευση και όχι επανεθνικοποίηση. Είναι μεγάλο το δίλημα και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά, διότι ε, έχουμε χώρες με συνδεδεμένες ε, ε, ενισχύσεις και εδώ φαίνονται τα αποτελέσματα. Ένας άλλος τομέας είναι τα δάση και αυτό το θίξατε. Κατά την τελευταία στρατηγική για τα δάση εργάστηκα κι εγώ και έρχομαι από μια περιοχή όπου ο τομέας της δασοκομείας παίζει μεγάλο ρόλο. Πιστεύω λοιπόν ότι το δάση είναι ο μεγάλος χαμένος στη μεγάλη αυτή συζήτηση για την προστασία του κλίματος και μόνο ένα ε, δάσος ε, που καλλιεργείται, που προστατεύεται ε, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης, ε, μόνο με σωστή πολιτική για τα δάση μπορούμε να έχουμε και σωστό σχεδιασμό. Ένα άλλο θέμα που με απασχολεί πολύ είναι η Συμφωνία Mercosur. Το παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυς, το γνωρίζω. Θα ήθελα να πω όμως ότι και ε, και στη ε, ε, Βολιβία έχουμε μεγάλο πρόβλημα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα δάση και όχι μόνο στην Βραζιλία. Το πρόβλημα της αποψήλωσης υπάρχει. Πρέπει λοιπόν να εφαρμοστούν εκεί πολιτικές που θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Και για τα υπόλοιπα θέματα συμφωνώ με τον προηγούμενο μιλητή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χόσλινγκ, ευχαριστούμε Υπουργέ που ήρθατε. Αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε και έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ε, μια αίσθηση business as usual ε, ότι ε, να αλλάξει λίγο η ΚΑΠ. Όχι, χρειάζεται ριζική αλλαγή. περιμένουμε να πάρουμε καινούρια δεδομένα. Εις ό,τι αφορά το κλίμα, το, κλίμα, το θέμα βιοπικιλότητας, εδώ οι προτάσεις Χόγκαν δεν μας δίνουν απαντήσεις και η δραματική αλλαγή του κλίματος έχει οξυνθεί κι άλλο. Ε, έχουμε πρόβλημα με τη συγκομιδή στη Γερμανία λόγω της μεγάλης ξηρασίας. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για τις λεπτομέρειες. 60% ε, στην πρώτη, στον πρώτο πυλώνα ε, μοιράζεται σε άμεσες πληρωμές και ε, εξακολουθούμε να δίνουμε ενίσχυση ανά εκτάριο και όχι με άλλα κριτήρια. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Νομίζω ότι δεν συμπεριλαμβάνομαι παρκώς το θέμα της βιοπικιλότητας. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Επίσης, ε, ε, για το Μερκοσούρ μιλήσατε κάπως ε, ασαφώς. Θα πρέπει να δούμε πολύ συγκεκριμένα τι γίνεται με τον περιορισμό της των εισαγωγών σόγιας και βοήου κρέατος ε, μετά από αυτά που γίνονται στη Βραζίλια. Πρέπει να δείξουμε σαφή ε, πολιτική. Δεν θα πρέπει να είμαστε γενικόλογοι στο θέμα της βιωσιμότητας, αλλαγής κλίματος κλπ. Ε, δεν μπορούμε να κάνουμε συμφωνίες με ανθρώπους ε, που ε, βάζουν οι ίδιοι φωτιές στα δάση τους και αυτό το επιτρέπει ο νόμος. για τα δάση, δεν, ε, αρκούν, δεν αρκεί μόνο η ε, σωστή ε, εκμετάλλευση των δασών για να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος. Χρειαζόμαστε και βιώσιμη πολιτική γιατί για τα δάση. Σε πολλές περιοχές ε, στην ε, Γερμανία έχουμε ε, προβλήματα με δάση από οξιές για παράδειγμα που δεν είναι πλέον βιώσιμες. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Τάβιτ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. στην Ανατολική Ευρώπη οι εργασιακές δομές στη Γεωργία είναι δυσμενείς για τους απασχολουμένους. Εκεί τι μέτρα θα λάβετε για να βελτιώσετε την κατάσταση. Δεύτερη ερώτηση. Πυρκαγιές στη Βραζιλία. Τι μηχανισμούς έχουμε για να βοηθήσουμε τη Βραζιλία να διορθώσει την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφο Γιώργη Γκίλ, εξ τη της συναδέλφου Μακιντάιρ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ε, α, παρακολουθώ την κοινή πολιτική εδώ και πολλά χρόνια και στο άρθρο 38 της Συνθήκης Λισαβόνας αναφέρονται οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινή πολιτική. Κατά τη γνώμη σας, δεν θα πρέπει να γίνει ένας απολογισμός ε, κατά πόσο έχουν υλοποιηθεί αυτοί οι στόχοι του άρθρου 38 της συνθήκης. Γιατί νομίζω ότι δεν έχουν ε, υλοποιηθεί αυτοί οι στόχοι ακόμη. Και θα πρέπει να κάνουμε πρώτα τον απολογισμό και κατά πόσο το νομοθετικό πακέτο θα συμβάλλει στην υλοποίηση αυτών των στόχων. Επίσης, ε, ε, μιλήσατε για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών αξιών, τα δικαιώματα του ανθρώπου και το κράτος δικαίου. Ε, έχουμε την θέση της Πολωνίας ε, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων και την περίπτωση αναστολής πληρωμών σε περίπτωση παραβίαση του κράτους δικαίου. Υπάρχουν όμως πολλές αφιβολίες για την κατάσταση αυτή. Σε πολλές περιπτώσεις η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση καταπατά τις συνθήκες. Ε, για παράδειγμα, η κινητοποίηση του άρθρου 7 κατά της Πολωνίας για, το, για την παραβίαση του κράτους δικαίου ε, ήταν απαράδεκτη και θα πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές και κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, δεν θα πρέπει να αφιερώσουμε κάποια κονδύλια της πολιτικής συνοχής για τη βελτίωση της ανάπτυξης της υπαίθρου. Συμφωνείτε με μια τέτοια πρόταση. Γιατί να μην αφιερώσουμε κονδύλια τη συνοχής για να στηρίξουμε τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φλάναγκαν. Δεν τον βλέπω όμως αυτή τη στιγμή. Ποιος θα μιλήσει εξ ονόματος της ΓΚΟΕ. Κανείς. Όχι. Δεν επιθυμείτε να λάβετε το λόγο. Υπουργέ. Τότε, Υπουργέ, θα μπορούσαμε να σας δώσουμε το λόγο για να απαντήσετε. Το πρώτο γύρο των απαντήσεων. Έχετε και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και για τις δύσκολες ερωτήσεις. Διαβλέπω το νόημά τους σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε. Στην ομιλία μου σας είπα ότι ήρθα να ακούσω τη γνώμη σας για τα σημαντικά αυτά θέματα και τις μεταρρυθμίσεις. Καταρχήν μερικές παρατηρήσεις. Χρειαζόμαστε γνήσια απλούστευση και η Φιλανδία προωθεί την απλούστευση εδώ. Δώσαμε μάχη για την απλοποίηση σε πολλές μεταρρυθμίσεις. Ε, και δεν ε, υλοποιήθηκαν όλες οι προτάσεις μας. Τώρα ήρθε η ώρα να πάρουν σάρκα και οστά. Προωθούμε πολύ την απλοποίηση και στην καθημερινή δουλειά των ε, γεωργών, των παραγωγών. Και έτσι θα υπάρξει και απλοποίηση σε διοικητικό επίπεδο επίσης, γιατί και αυτό το θέλουμε. Πολλά ακούστηκαν για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ γι' αυτό. Ένα σημαντικό κομμάτι στο πλαίσιο του πολιετούς πλαισίου είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων και αυτών που χρηματοδοτούμε. Αυτή είναι και η γραμμή της Φιλανδίας. Αυτό το λέω ως εκπρόσωπος της Προεδρίας. Το έχω επαναλάβει πολλές φορές και δημοσίως και στο Συμβούλιο. Δεν μπορούμε να έχουμε αυξανόμενες απαιτήσει και λιγότερες πληρωμές. Αυτή δεν είναι εξίσωση λειτουργική. Πρέπει να υπάρχει ένα ισορροπημένο πλαίσιο στο πολιετές πλαίσιο. Οι περικοπές στον δεύτερο πυλώνα είναι μεγαλύτερες από ό,τι στον πρώτο. Πρέπει να το δούμε αυτό πιο προσεκτικά. Για το δεύτερο πυλώνα μπορέσαμε σε πολλά κράτη-μέλη να δημιουργήσουμε συστήματα που προσφέρουν κίνητρα σε πολλούς εμπλεκομένους και πολλοί παραγωγοί ε, θέλουν. Και βεβαίω πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τι διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Πρέπει αυτέ να τις λάβουμε περισσότερο υπόψη εδώ και όχι στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα. Αλλά η ισορροπία, η ευθυδικία, η δικαιοσύνη είναι σημαντικά στις πολιτικές μας. Τα θέματα της χρηματοδότησης είναι, όπως είπα, μεταξύ των προτεραιοτήτων της Φιλανδικής Προεδρίας. Προς ασφαλώς, ασφαλώς το Brexit δημιουργεί κάποια ανασφάλεια για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρέπει να το θεωρήσουμε ως δεδομένο αυτό στις ε, προετοιμασίες μας. Γιατί έχουμε κάνει προετοιμασίες ε, και εξετάσαμε διάφορα σενάρια για το Brexit. Ε, δηλαδή το Brexit και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Υπάρχουν λοιπόν σενάρια, εναλλακτικές ε, εργασίες που έχουν γίνει. Και θα προχωρήσουμε ανάλογα με το σενάριο που θα διαμορφωθεί. Τώρα, η δασική πολιτική είναι πολύ σημαντική και η μεταρρύθμισή της είναι επίσης σημαντική. Ε, εγώ ε, μεγάλωσα στα δάση, έχω παρελθόν που είναι συνδεδεμένο με αυτά. Το 70% της ε, έκτασης της ε, Φιλανδίας καλύπτεται από δάση. Ξέρω πολλά για τα δάση. Πριν περάσουμε σε θέματα στρατηγικής, θα ήθελα να πω ότι μπορούμε και πρέπει να δράσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να λάβουμε υπόψη μας όλα τα διαφορετικά προβλήματα των δασών, αφού τα δάση ε, είναι πολύ σημαντικά για την παγίδευση του άνθρακα. Ε, όσο περισσότερα δάση, τόσο μεγαλύτερη η παγίδευση του άνθρακα. Είναι νόμος της φύσης. Ό,τι είναι πράσινο παγιδεύει τον άνθρακα και τα δάση είναι πράσινα. Και αυτό το θέμα έχει τεράστια σημασία. Και σίγουρα όταν ε, χρησιμοποιούμε τα δάση με βιώσιμο και ε, ορθολογικό τρόπο ε, μπορούμε να έχουμε προϊόντα που θα αντιμετωπίσουν την μια ανανεώσιμη ενέργεια. Ε, εμείς θέλουμε να γίνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ουδέτεροι από άποψη χρήσης άνθρακα και θέλουμε να έχουμε μηδενικές εκπομπές στη περιφέρεια της Ένωσης. Ε, δεν ε, μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε με τις μη ανανεώσιμες. Πρέπει να εισαγάγουμε την κυκλική οικονομία, βιώσιμο, βιώσιμη αντιμετώπιση των δασών και Θέλουμε μέσω της πολιτικής των δασών να διασφαλίσουμε και την βιοπικιλότητα. Ε, πολλά, πολλοί στόχοι μπορούν να επιτευχθούν εδώ μαζί, στα πλαίσια της ίδιας πολιτικής. Ε, γι' αυτό είναι σημαντικά τα δάση. Και Επίσης είναι και μεγάλο τεράστιο οικονομικό κεφάλαιο τα δάση, υπό πολλές έννοιες. Η αναβάθμιση της, για τα, της πολιτικής για τα δάση μετά το 2020 είναι ο στόχος μας και ο τομέας των δασών θα είναι τομέας κέρδιας σημασίας για να βελτιώσουμε την βιοοικονομία μας, την ανταγωνιστικότητά μας και για να προσφέρουμε νέες ευκαιρίες στον αγροτικό κόσμο. Τον Απρίλιο το Συμβούλιο απευθύνθηκε στην Κομισιόν για μια καλύτερη δασική πολιτική από άποψη περιβαλλοντική και βιοοικονομική. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη χρήση των δασών όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά διεθνώς, παγκοσμίως. Ως προεδρία, προεδρεύουσα χώρα, η Φιλανδία θέλει να δώσει μια ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων επί αυτών των θεμάτων στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου, όπου έχουμε δύο συζητήσεις. Η πρώτη συζήτηση έγινε ήδη στην αρχή Ιουλίου. Έγινε στο Ελσίνκι μια μεγάλη ε, διάσκεψη για την βιοοικονομία με ε, πολλούς συνέδρους και επίσης ε, θα γίνει και μια ε, εκδήλωση με τους επικεφαλείς των τομέων και διευθύνσεων δασικής πολιτικής. Μια άλλη ερώτηση αφορούσε το αν μπορούμε να επιτύχουμε στόχους της ΚΑΠ αν δώσουμε περισσότερες εξουσίες στα κράτη-μέλη. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αναπτύξουμε το σύστημα όπως το πρότεινε η Κομισιόν, ούτως ώστε να έχουμε στρατηγικά ε, προγράμματα που θα υποβάλλονται από τα κράτη-μέλη, θα εξετάζονται από, και θα αξιολογούνται από την Κομισιόν, ούτως ώστε ο στρατηγικός στόχος που έχει τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εφαρμόζεται. Έτσι πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα. Συμφωνώ απόλυτα με τους ομιλητές που είπαν ότι η παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Και θα έλεγα ότι είναι, είναι το επίκεντρο της ΚΑΠ, ο κεντρικός άξονας, όλα γυρίζουν γύρω από αυτόν. Η Γεωργία αυτό το σκοπό έχει την παραγωγή τροφίμων. Ε, συμμερίζομαι τις ανησυχίες για την Βραζιλία, τη Βολιβία και πολλά άλλα μέρη του κόσμου όπου τα δάση καίγονται. Αυτό μας πάει πίσω, δεν βοηθάει καθόλου. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις πυρκαγιές, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να τις προλαμβάνουμε τις δασικές πυρκαγιές. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές κάθε κράτους μέλους. Πρέπει να υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ κρατών για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Είναι αλήθεια ότι τώρα ε, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στη Βραζιλία αλλά το πρόβλημα παρουσιάζεται και σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου. Επίσης ακούσαμε ότι χρειάζονται πολύ ριζοσπαστικές αλλαγές για να ε, εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις και οι στόχοι μας. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι είμαστε ένας διεθνός παίκτη στις διεθνείς αγορές. Ε, θα πρέπει να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, ε, σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που σχεδιάζουμε τώρα και που έχει προχωρήσει αποτελεί μια λύση. Δηλαδή θα επιτύχουμε μια αλλαγή που τη θέλουμε όλοι και θα είναι βιώσιμη και οικονομικά και κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Αυτό είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι μετριέται η βιωσιμότητα των δράσεων. Τώρα η Συμφωνία Μερκοσούρ είναι μια συμφωνία ε, απαιτητική. Ε, θέτει περιορισμούς, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται. Δεν γίνεται διαφορετικά δεν μπορούμε να υπογράφουμε συμφωνίες με κάθε κόστος. Θα πρέπει να παρακολουθούνται, θα πρέπει να τηρούνται, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι συμφωνίες. Επίσης, ε, ε, θέσατε και κάποια ζητήματα που δεν είναι στο, υπό τη δική μου ευθύνη. Θα ήθελα όμως να κάνω κάποια σχόλια παρόλα αυτά η κατάσταση των γεωργών. Εξίσου δύσκολη είναι η κατάσταση για τους παραγωγούς. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί συνολικά η κατάσταση ε, στη γεωργία και να λειτουργούν με σωστά οι ε, αγορές. Εδώ το Κοινοβούλιο έκανε εξαιρετική δουλειά. Σας ευχαριστώ και ε, πραγματικά συμβάλλατε στο να έχουμε ε, ε, αγορές δίκαιες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για κερδοφόρο παραγωγή. Η κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να δίνει κίνητρα για κερδοφόρο γεωργική παραγωγή. Και για να ολοκληρώσω, πώς ε, αξιολογείται η ΚΑΠ. Εμείς ε, αξιολογούμε τις προτάσεις για μεταρρυθμίσεις στην ΚΑΠ και θα συμπεριλάβουμε πολλά θέματα, όπως να παρακολουθούμε τι... τα επιτεύγματά μας, τα αποτελέσματα. Τώρα, για τα μεγάλα αρπακτικά ζώα, λύκοι, αρκούδες κλπ. Όλοι περιμένουμε από το δικαστήριο ε, αποφάσεις και ο στόχος μας είναι τα κράτη-μέλη να έχουν με τον α ή β τρόπο να, ε, την εξουσία για να ε, λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τα μεγάλα ζώα και να προλαμβάνουν του τα, τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Όταν λάβουμε την απόφαση του δικαστηρίου θα προχωρήσουμε σε στις λεπτομέρειες και τότε η ε, Κομισιόν θα σχεδιάσει το δικό της πρόγραμμα. Τότε θα έρθει η ώρα για να συζητήσουμε τις συγκεκριμένες μεθόδους. Σίγουρα τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία για να αντιμετωπίζουν για, ε, ε τα, τους κινδύνους στα μεγάλα αυτά ζώα. αυτή είναι η εμπειρία από τη Φιλανδία. Ξέρω ότι υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης μεγάλα προβλήματα. Έχουμε ακούσει παρόμοια προβλήματα και από εσά. Αναγνωρίζω ότι είναι ε, ένα θέμα έχει εντοπιστεί, είναι στην ημερήσια διάταξή μας και θα παραμείνει. Με ευχαριστώ πολύ ε, για τις απαντήσεις αυτές. Και τώρα προχωρούμε στους επόμενους ομιλητές. Πάμε καλά από χρόνο και θα πρότεινα να γίνει πινκ-πονγκ, ερώτηση-απάντηση η συζήτηση. Μετά την ερώτηση του βουλευτή, της ε, βουλευτή, να απαντάει αμέσως ο Υπουργός. Η κυρία Σχρέιρ Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, συγχαρητήρια προς τον Υπουργό. Προηγουμένως, ε, σας είδα και στην Επιτροπή Αλίας ε, πολύ σημαντικό εδώ αυτό που λέτε, εκτός από την κλιματική αλλαγή και τη Συμφωνία για το Κλίμα, έχουμε και παραγωγή τροφίμων και ασφάλεια τροφίμων. Εδώ είμαστε στην Επιτροπή Γεωργίας και το ξέρουμε αυτό, αλλά στις άλλες επιτροπές κυριαρχεί συνήθω το κλίμα και τα άλλα είναι υποδέστερα. Πώς σκέφτεστε ε, να διατηρήσετε την παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη και την παραμονή των νέων αγροτών στη Γεωργία. Δεύτερον, Δύο μέρες ήμουνα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, ΙΝΤΑ, και εκεί συζητάμε και θέματα Μερκοσούρ και έπονται ε, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Υπάρχουν άλλοι τομείς που είναι πιο σημαντικοί από τη Γεωργία, αλλά πραγματικά κοιτάξτε τους αριθμούς ε, ε, ε, και να υπάρχουν πραγματικά αποζημιώσεις για τους ε, δικούς μας αγρότες. Τι θα γίνει με αυτό. Και ένα τρίτο πολύ σημαντικό, το οποίο αναφέρατε και εσείς για το λύκο, συγχαρητήρια για το όσα λέτε, στις διακοπές άκουσα από ένα καθηγητή ότι δεν υπάρχει ο πραγματικός λύκος, ότι είναι όλα υβρίδια ε, και τα οποία μπορούμε να κυνηγάμε άφοβα. Δεν υπάρχει 100% λύκος. Αλλά το θέμα της αντοχής στα αντιβιωτικά επίσης με ε, απασχολεί πάρα πολύ. Το είχαμε δει και στην περιεργόμενη θητεία. Εμείς έχουμε προχωρήσει πολύ, αλλά δεν έχουν προχωρήσει καλά ακόμα στις, ε, στους ελέγχους όλα τα κράτη-μέλη. Εσείς πώς θα το φροντίσετε αυτό και πώς θα το ρυθμίσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, παρακαλώ να απαντήσετε. Απάντηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους βουλευτές ε, για τις ερωτήσεις. Ε, συμφωνώ πολύ με αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η παραγωγή τροφίμων είναι ε, κομβικό στοιχείο και συστατικό ε, της ευημερίας μας αλλά και της ίδιας μας τη ζωή στην Ευρώπη. Αν δούμε τη δημογραφική πρόγνωση, καταλαβαίνουμε ότι τα τρόφιμα και η παραγωγή τροφίμων δεν είναι κάτι το αυτονόητο και το προφανές. Χρειάζονται δουλειά. Συνέχεια. Η παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να είναι και βιώσιμη φυσικά, αλλά χρειάζεται δουλειά. Μιλήσατε για τους νέους αγρότες. Και εγώ ανησυχώ αν δούμε τις στατιστικές για τη μέση ηλικία των αγροτών και πώς αυτή εξελίσσεται, προφανώς γυράσκουν και οι αγρότες συνεχώς. Και αν θέλουμε να ε, εισάγουμε νέες τεχνολογίες και στη γεωργία, είναι προφανές ότι οι νέοι είναι πιο πρόθυμοι και ε, ε, θέλουν να υιοθετήσουν αυτές τις τεχνολογίες. Βέβαια και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πολίτε ε, διστάζουν, προχωρούν και αυτοί στις νέες τεχνολογίες. Αλλά αν οι νέοι χάσουν την πίστη τους στη γεωργία, ε, δεν πρόκειται να ασχοληθούν με τη γεωργία. Δεν θα γίνουν αγρότες και παραγωγοί τροφίμων. Θα ασχοληθούν με κάτι άλλο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουν προοπτικές από τη γεωργία και οι νέοι και να κατανοούν ότι η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων είναι κάτι το ελκυστικό και ότι έχουν μέλλον σε αυτή τη δραστηριότητα. Μιλήσατε για τους λύκους υβρίδια. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε ε, αυτό το φαινόμενο να ε, διασταυρώνονται με σκύλους και να ε, γεμίζει ύπεθρος ε, λύκους ε, που είναι διασταυρωμένοι σκύλους, λυκόσκυλα ουσιαστικά και δεν είναι γνήσιοι λύκοι. Επίσης, οι λύκοι, όπως και τα ζώα γενικά, δεν γνωρίζουν σύνορα, ούτε διαβατήρια, ούτε διατυπώσεις στα σύνορα. Δύο λόγια τώρα για τη γεωργία και το εμπόριο και τις εμπορικές συμφωνίες. Φυσικά όλες οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ισορροπία και όλες οι συμφωνίες. Η ισορροπία αυτή είναι εξαιρετική σημασία. Υπάρχουν κάποια ευαίσθητα προϊόντα ε, τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Και φυσικά θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε ποσοστώσεις. Και όρια στις εισαγωγές και τα και θα πρέπει να είμαστε πάντα πολύ προσεκτικοί όταν διαπραγματευόμαστε εμπορικές συμφωνίες. Συμφωνώ πολύ τους λοιπόν. Επίσης για την αντοχή των μικροβίων στα αντιβιωτικά είναι τεράστιο πρόβλημα το οποίο θα ενταθεί ακόμα περισσότερο και συνιστά παγκόσμια απειλή. Θυμηθείτε τι έγινε πριν από δύο χρόνια στο Παγκόσμιο Φόρουμ όταν η Υπουργοί Γεωργίας 100 χωρών ε, συζητούσαν αυτό το θέμα. Και αυτό ήταν το βασικό μας ε, μέλημα. Δεν είναι πρόβλημα μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι παγκόσμιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. <laughs> Δεν λειτουργεί πολύ καλά αυτό το σύστημα με το ping-pong. Ερώτηση-απάντηση από χρόνο και τήρηση του χρόνου. Οπότε πάμε πάλι στην παραδοσιακή μέθοδο. Επιστρέφουμε. Ένα λεπτό κάθε ομιλητής και ο Υπουργός στο τέλος για να απαντήσει. Και αν έχουμε χρόνο, από εκεί και πέρα μπορεί να γίνουν και συμπραγματικέ ερωτήσεις και διευκρινιστικές. Νομίζω είναι καλύτερη αυτή η λύση. Παρακαλώ να με συμπαθάτε. Και εγώ μαθαίνω τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Ήθελα να κάνω λίγο πιο ζωηρή τη συζήτηση. Ε, συνάδελφος ε, ε, Αφράμ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις. Φέτος, για πρώτη φορά, το Συμβούλιο ανήγγειλε ότι δεν θα ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μέχρι ότου ξεκαθαρίσει η εικόνα του πλαισίου του ΠΔΠ. Μπορείτε να μας ε, δώσετε ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τις συζητήσεις αυτές. Επίσης, 10 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό που προτείνεται για τη γεωρική έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε ό,τι αφορά τη γεωρική έρευνα μεταξύ των κρατών μελών. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια λύση ώστε τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων ε, να είναι ανοιχτά σε όλα τα κράτη-μέλη, ακόμη και σε εκείνα που δεν έχουν τόσο προηγμένη γεωργική έρευνα. Ευχαριστώ κύριε Σαντέρ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, όλοι θέλουμε να προαγάγουμε μια γεωργία που θα παρακολουθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τις περιβαλλοντικές αλλαγές και τις κλιματικές αλλαγές. Και φυσικά έχουμε αναπτύξει κάποια οικολογικά προγράμματα και είμαστε υπέρ μιας ε, ισχυρής αιρεσιμότητας. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες ε, πληροφορίες για τις συζητήσεις και την πορεία των συζητήσεων για τα θέματα αυτά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε για να αποφύγουμε τις στρεβλώσεις ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φροντίσουμε η κοινή γεωργική πολιτική να, γίνει, να μείνει πραγματικά κοινή και ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική. Και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέσει κάποια όρια, ανώτατα και εκατότατα, για να πλαισιώσουμε καλύτερα τα κονδύλια του πρώτου ή του δεύτερου πυλώνα. Μπορείτε να μας δώσετε πιο διεξοδικές πληροφορίες για την πορεία των συζητήσεων και για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, και εγώ γεννήθηκα σε, στα δάση, όχι όμως στην ελεύθερη Φιλανδία, αλλά στη Σιβηρία, εκεί που είχαν εξοριστεί οι γονείς και παππούδες μου. Και τα δάση της Σιβηρίας α, ε, μαστίζονται από πυρκαγιές, όπως και τα δάση της Βραζιλίας. Ε, αναφέρατε την στρατηγική για τα δάση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να προστατεύσουμε τα δάση και να περιορίσουμε την παρακμή τους. Μην ξεχνούμε ότι τα δάση είναι οι πνεύμονες ε, της Ευρώπης και του κόσμου. Επίσης, ε, μιλήσαμε για ισορροπημένο και θεμητό ανταγωνισμό. Πώς λοιπόν θα αποτρέψουμε τις άδικες ενισχύσεις, άδικες ε, πληρωμές, γιατί οι γεωργοί στη Λιθουανία και στι βαλτικέ χώρε λαμβάνουν πολύ χαμηλότερε ενισχύσει. Πρέπει να υλοποιήσουμε μια εξίσωση ε, των ενισχύσεων, όπως είπαμε, μέχρι το 2020. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για την ομιλία σας. Συμφωνούμε ότι δεν μπορούμε να οριστικοποιήσουμε την κοινή γεωρική πολιτική και τη μεταρρυθμισή της πριν ε, την προηγούμενη απόφαση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί είναι αλληλένδετα τα δύο θέματα. Είμαι ευρωβουλευτής από την Ουγγαρία. Θα πρέπει πρώτα λοιπόν να δούμε τα αριθμητικά στοιχεία και μετά να αποφασίσουμε για τα κονδύλια της κοινή γεωργικής πολιτικής. Στο Κοινοβούλιο επίσης και στην Επιτροπή Γεωργίας θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα στηρίξουμε το ισχύον πλαίσιο της ΚΑΠ ή θα ξεκινήσουμε την όλη διαδικασία εκ του μηδενός. Είναι σημαντικό να λάβουμε τη σχετική απόφαση. Επίσης, ας μην ξεχνούμε ότι η γεωργή σε τελική ανάλυση και κυρίως οι μικρομεσαίοι αγρότες, ε, οι οικογενικές εκμεταλλεύσεις ε, ε, είναι οι, αυτοί που θα επηρεαστούν κυρίως από τις προτεραιότητες και τη διάρθρωση της μελλοντική ΚΑΠ. Θα πρέπει να καταστήσουμε την ΚΑΠ προβλέψιμη για να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να προγραμματίσουν το μέλλον τους. Αν δεν λυθεί τελικά απόφαση, έγκαιρη απόφαση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, τι σκοπεύει να κάνει η Φιλανδική Προεδρία για τη μεταρρυθμίση της ΚΑΠ. Θα την αναβάλει. Τι κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να γίνει αν δεν λυθεί εγκαίρως απόφαση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κυρία Κατάινεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Τα σχόλιά σας είναι πιστικά, ε, συνεκτικά και συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στα βασικά που είναι η παραγωγή τροφίμων στην ΚΑΠ και ε, πρέπει τα τρόφιμα να είναι εξασφαλισμένα παντού στην Ευρώπη. Ε, η ε, σήμανση προέλευσης είναι πολύ σημαντική. Έχουμε ένα πιλωτικό έργο στη Φιλανδία, σύμφωνα με το οποίο τα εστιατόρια πρέπει να έχουν σήμανση για το κρέας, για την προέλευση. Είναι σημαντικό αυτό για την υγεία, για την ασφάλεια των τροφίμων. Καλό θα ήταν παρόμοια νομοθεσία να υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να ξέρουν τι τρώνε και μακροπρόθεσμα θα πρέπει αυτή η νομοθεσία να καλύψει και όλα τα βασικά γεωργικά προϊόντα, ώστε οι καταναλωτές να αποφασίζουν ήδη αν θέλουν να φάνε τρόφιμα από κοντινές περιοχές ή από μακρινές περιοχές. Ε, η ερώτησή μου είναι λοιπόν τι θα κάνει το Συμβούλιο σχετικά με τη σήμανση της προέλευσης των προϊόντων επί Φιλανδικής Προεδρίας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ροπή. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή που μας δίνετε να, σας, ε, να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων. Ε, χάρηκα που είπατε ότι το πιο σημαντικό ε, για την Προεδρία σας είναι οι κανόνες της ΚΑΠ. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε ε, πολλές γνώμες πάνω σε αυτό το θέμα. Ελπίζω να καταλήξουμε σε κοινό παρονομαστή. Και ελπίζω να ολοκληρωθεί και η διαβούλευση και να αποφασιστεί το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλιώς δεν γίνεται. Είναι σημαντική η ανταγωνιστικότητα. Οι διαφορές στις πληρωμές μεταξύ χωρών είναι μεγάλες. Πολλές φορές είναι διπλάσιες ή τριπλάσιες. Ε, έτσι μπαίνει θέμα ανταγωνιστικότητας ε, στις κοινέ αγορές. Η γεωργική παραγωγή λοιπόν μειώνεται στις βαλτικές χώρες και είναι πολύ λυπηρό να βλέπουμε Ιστονούς, Λετονούς ε, να πηγαίνουν στη Δανία για να ασχοληθούν με τη γεωργία που θα μπορούσαν να το κάνουν στη χώρα τους, μένοντας στην περιοχή τους και μαζί με τις οικογένειές τους. Ερωτώ λοιπόν, ποια είναι η θέση σας σχετικά με την εξωτερική σύγκληση και πότε θα πρέπει να περιμένουμε τις σχετικές αποφάσεις που είχαν ληφθεί από το Συμβούλιο πριν από 15 χρόνια ώστε ε, το 2013 να φτάσουμε σε ένα ε, μέσο όρο παντού. Αυτό δεν έχει γίνει. Κάτι άλλο, οι πληρωμές ε, προς τους αγρότες. Οι αγρότες δεν έχουν μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη, αυτό είναι γνωστό. Και οι τιμές αγοράς είναι πολύ χαμηλές σε πολλές περιοχές. Τι θέση έχετε για τις δίκαιες πληρωμές και δίκαιες ε, τιμές αγοράς για τους αγρότες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίαση. Την ίδια ερώτηση έχω και εγώ σχετικά με την διαδικασία σύγκλησης των άμεσων πληρωμών είμαι από ένα κράτος μέλος που παίρνει πολύ λιγότερες ε, επιδοτήσεις από άλλες. Όταν μιλάμε για ευθυδικία και δικαιοσύνη πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό. Γιατί όλοι λειτουργούμε στην ίδια ενιαία αγορά. Είναι δίκαιο και σωστό όλοι οι Ευρωπαίοι αγρότες λοιπόν να ωφελούνται από τις ίδιες προϋποθέσεις εις ό,τι αφορά τις γεωργικές επιδοτήσεις. Δεύτερον, κυρία Υπουργέ, μιλήσατε θετικά για τη Συμφωνία Μερκοσούρ. Όμως θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε πραγματικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρκετούς μηχανισμούς για να διασφαλίσει ότι η περιφέρεια της Ένωσης δεν θα κατακλειστεί από προϊόντα διαφορετικών προτύπων από τα ευρωπαϊκά. Πού αναφέρομαι συγκεκριμένα. Σήμερα οι χώρες του Μερκοσούρ χρησιμοποιούν 74 ζυζανιοκτώνα και εντομοκτώνα που απαγορεύονται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να τους σταματήσουμε από την πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αλλιώς θα δυσκολέψουν τα πράγματα ακόμη περισσότερο για τους δικούς μας τους αγρότες που θα υπομισθούν μεγαλύτερο κόστος και θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρότερους κανόνες. Ενώ από την άλλη πλευρά δεν έχει νόημα να μιλάμε για τη μικροβιακή αντοχή αν αναγκάζουμε μόνο τους δικούς μας τους γεωργούς να σέβονται αυτές τις αρχές ενώ ανοίγουμε διάπλατα τις πόρτες μας σε αγρότες που δεν είναι υποχρεωμένοι να ε, ακολουθούν αυτές, αυτούς τους περιορισμούς. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Κύριε Γιλάρ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που μας παρουσιάσατε τις προτεραιότητες της Φιλανδικής Προεδρίας στη Γεωργία. Θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημαντικά θέματα που ελπίζω να απασχολήσουν και την Προεδρία. Καταρχήν, ισορροπία των εμπορικών συμφωνιών που πλήττουν κυρίως στην Μεσογειακή Γεωργία. Δεύτερον, τα μεσογειακά προϊόντα είναι ευαίσθητα και τα σπεριδοειδή και το ρύζι είναι αυτά που περισσότερο έχουν πληγεί. Σε ό,τι αφορά τη στήριξη της καινοτομία στη Γεωργία, τι σκοπεύει να, να προτείνει η Φιλανδική Προεδρία για τις νέες τεχνικές βελτίωσεις, new breeding techniques και τι γίνεται με την αναθεώρηση της οδηγίας για τους σπόρους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Λεμπρετών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπουργέ, θέλετε να εξασφαλίσετε τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία της γεωργίας σε όλα τα κράτη-μέλη. Θετικό είναι αυτό το μήνυμα που στέλνετε στους αγρότες μας. Παράλληλα όμως, μόλις υποστηρίξατε τη συμφωνία με τις χώρες Mercosur. Όμως αυτή η συμφωνία κινδυνεύει να κατακλείσει με φτηνά προϊόντα τις αγορές μας που παράγουν οι γεωργικοί γίγαντες όπως είναι η Βραζιλία ή η Αργεντινή. Οι Γάλλοι αγρότες ανησυχούν έντονα και το δήλωσαν το καλοκαίρι και μάλιστα ε, με τρόπο έτσι θορυβόδη και επιτέθηκαν σε γραφεία Γάλλων βουλευτών. Πώς συνάδουν αυτές οι δύο επιθυμίες σας, δηλαδή από τη μια να είναι η κερδοφόρα η Γεωργία και από την άλλη να υποστηρίζετε την συμφωνία Μερκοσούρ που ε, απειλεί το εισόδημά τους. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα πρότεινα να περάσουμε σε ένα γύρο απαντήσεων και στη συνέχεια οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Παρακαλώ, Υπουργέ. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Θα α, ε, ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας και για τις ερωτήσεις σας. Ε, ρωτάτε αν ισχύει ότι η κοινή γεωργική πολιτική ε, δεν πρόκειται να προχωρήσει αν δεν προχωρήσει το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ισχύει αυτό και είναι επόμενο και φυσικό. Χρειαζόμαστε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε την ε, μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αν βάλουμε 10 ε, δισεκατομμύρια για την έρευνα εκεί. Από εκεί και πέρα τι θα τα κάνουμε αυτά τα αποτελέσματα. Μα χρειαζόμαστε έρευνα και μελέτες για να φτάσουμε στους στόχους που έχουμε θέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ε, τα χρήματα αυτά για την έρευνα. Είναι πολύ σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάλογα με τις συνθήκες χρειαζόμαστε την έρευνα. Είναι σημαντικό στοιχείο η έρευνα. Είναι γεγονός αυτό. Επίσης, η γεωργία θα πρέπει να είναι βιώσιμη και ως προς το κλίμα και την κλιματική αλλαγή. Χρειαζόμαστε μια κοινή γεωργική πολιτική για να μπορέσουμε να φτάσουμε στους στόχους μας. Για την πολιτική των δασών. Είναι πολύ σημαντικό φυσικά να προστατεύουμε τα δάση μας. Δεν γνωρίζουν όλοι τα της δασοκομείας. Ε, σε όλες τις χώρες υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν από δάση ε, και οι στόχοι μπορεί να είναι διαφορετικοί από χώρα σε χώρα, αλλά ταυτόχρονα να επιδιώκουμε διάφορους στόχους. Ε, για το χρονοδιάγραμμα που ρωτήσατε, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι σαφές και το επαναλαμβάνω ξανά. Είναι μέγα ζήτημα αυτό για τη δική μας Προεδρία. Πραγματικά θέλουμε να το προωθήσουμε και να επιτευχθεί πρόοδος και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα το συζητήσει τον Οκτώβριο. Από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Θα δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ο καθένας στον τομέα του θα υπάρξει λύση από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Θα δούμε τι θα γίνει και με τις πληρωμές και κυρίως τις γεωργικές πληρωμές. Ε, αυτό είναι επίσης ε, τμήμα του πακέτου των πολιετών δημοσιονομικών ε, προοπτικών και του πλαισίου. Φυσικά, εάν υπάρξουν καθυστερήσει, θα συνεχιστεί η μεταβατική περίοδο, θα παραταθεί. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν οι μακρέ ε, μεταβατικέ περίοδοι, γιατί προκαλούν παντού ανασφάλεια. Όχι μόνο στου αγρότε, σε όλου του τομεί. Και είναι πολύ σημαντική η έννοια της σταθερότητας για τους αγρότες. Το έχω τονίσει αυτό. Βεβαίω θα πρέπει να παίρνουμε αποφάσει με προσοχή και όχι βεβαιασμένα, αλλά κάποια στιγμή να προχωράμε κιόλα. Σε ό,τι αφορά τι ετικέτε προέλευση, σήμανση, ε, χαίρομαι για το σχόλιο αυτό που κάνατε. Όταν ρωτούμε τους Ευρωπαίους καταναλωτές εάν ε, τους ενδιαφέρει η προέλευση των τροφίμων που καταναλώνουν, μας απαντούν ότι βεβαίως και ενδιαφέρονται. Θέλουν να γνωρίζουν ε, οι καταναλωτές και θέλουν καλύτερη σήμανση των προϊόντων ως προς την προέλευση. Προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε. Βεβαίως την τελική επιλογή την έχει πάντα ο καταναλωτής και θα πρέπει να γνωρίζει. Υπάρχουν ελλείψεις στην νομοθεσία για τη σήμανση της προέλευσης. Αυτό το συζητούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και καιρό και πριν αναλάβουμε την Προεδρία μάλιστα. Σας απαντώ λοιπόν ότι βεβαίως θέλουμε να ε, προωθήσουμε και αυτό το θέμα τη σήμανση της προέλευσης των προϊόντων για να λειτουργεί σωστά η εσωτερική αγορά. Ρωτήσατε για πιο δίκαιες αγορές τροφίμων. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό στοιχείο η δικαιοσύνη και θα ασχοληθούμε και με αυτό το ζήτημα. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο ε, το Κοινοβούλιο ασχολήθηκε με αυτό το θέμα και πραγματικά πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προεργασία που έχει γίνει. Είναι σαφές Γιατί και αυτό ανήκει στη βιώσιμη γεωργία και τη βιώσιμη γεωργική παραγωγή. Είναι βασική προϋπόθεση και προαπαιτούμενο για μια βιώσιμη κερδοφορία της γεωργίας. Για ποιο λόγο. Διότι το σύστημα πληρωμών δεν παρακολουθεί το κόστος. Το σύστημα πληρωμών είναι αποτέλεσμα πολιτικών διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει όμως ε, να δούμε τι γίνεται και με την εξέλιξη του κόστους παραγωγής που αντιμετωπίζει ο παραγωγός και το επομίζεται. Θα πρέπει οι ενισχύσεις και οι πληρωμές και οι επιδοτήσεις να λαμβάνουν υπόψη ε, το κόστος, ε, γιατί συνεχώς διευρύνεται η ψαλίδα. Κάτι ρωτήσατε για το Μερκοσούρ και πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι εμπορικές συμφωνίες δεν θα επιτρέψουν ε, την κυκλοφορία απαγορευμένων προϊόντων στην αγορά. Χρειαζόμαστε μηχανισμούς φυσικά ε, πρόληψης ε, κυκλοφορίας ανεπιθύμητων προϊόντων και εισαγωγής τους. Θα πρέπει να συνεχίσουμε και εκεί την προσπάθειά μας. Αναφερθήκατε στις νέες τεχνολογίες και τεχνικές βελτίωσης ε, breeding techniques. Έχουμε την ΕΦΣΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας ε, Τροφίμων, που κάνει τις αξιολογήσεις συνεχώς και τις μελέτες και εμπιστευόμαστε τον οργανισμό αυτό. Ε, σε πολλούς τομείς έχουμε εξελίξεις και στη γεωργία ε, τεχνολογικές και θα πρέπει κάθε φορά να μελετούμε ε, αυτά τα θέματα και από την σκοπιά που λέει ότι δεν θέλουμε να μείνουμε πίσω στις εξέλιξεις. Χρειαζόμαστε τις νέες τεχνολογίες, τις νέες βιώσιμες μεθόδους για να μπορούμε να λειτουργούμε και στη γεωργία. Και φυσικά θα πρέπει κάθε φορά να αξιολογούνται ε, με ένα ε, κριτικό ε, βλέμμα και οι καινοτομίε, αλλά χρειάζονται και οι καινοτομίε. Και ένα ακόμα σχόλιο που είχε να κάνει με την μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τους σπόρους, για το πολλαπλασιαστικό υλικό. Ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες ε, υποθέσεις και επιθυμίες να ενισχυθεί αυτή η νομοθεσία. Ελπίζω και στο νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βρει αντανάκλαση αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για τις διεξοδικές απαντήσεις. Πάμε τώρα στον επόμενο γύρο, ο συνάδελφος Τεσέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και εσάς κύριε Υπουργέ για το χρόνο που μας αφιερώνετε σήμερα. Όπως ακούσαμε σήμερα, μόνο 6% των ε, Ευρωπαίων γεωργών είναι κάτω των 35 ετών. Η γεωργική δημογραφία μας προβληματίζει ιδιαίτερως και θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων και για την μεταρρυθμίση της ΚΑΠ, ώστε το μέλλον της γεωργίας να επιστρέψει στους νέους, γιατί σε αυτούς ανήκει. Αναφερθήκαμε και στο θέμα των λύκων και δεν θα πρέπει στο μέλλον το είδος ε, που χρήζει προστασίας να είναι οι ίδιοι γεωργοί και να απειλούνται οι ίδιοι γεωργοί από εξαφάνιση. Κύριε Υπουργέ, πολύ αναφέρθηκα στο θέμα αυτό και είναι σημαντικό ε, και σας προβληματίζει και εσάς να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της γεωργίας. Βέβαια, πέραν των φιλοδοξιών μας, το διακύβευμα είναι κυρίως ευρωπαϊκό και θα πρέπει να διαρωτηθούμε τι μέτρα μπορούμε να εφαρμόσουμε για να επιτύχουμε την ηλικιακή ανανέωση στη Γεωργία και μάλιστα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί αυτό το θέμα μας είναι προσφυλές. Τι συγκεκριμένες δράσεις σκοπεύετε να αναλάβετε για να προσελκύσετε νέους στη Γεωργία σε όλα τα κράτη-μέλη και να επιτύχουμε έτσι την ηλικιακή ανανέωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα λίγο να επανέλθω στο Brexit, που είναι από τα πιο επίγοντα θέματα της Προεδρίας σας. Δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει τέλη Οκτωβρίου, αλλά πραγματικά ε, πιστεύω ότι θα φύγουν οι Βρετανοί. Το Brexit λοιπόν θα έχει επιπτώσεις όχι μόνο στον προϋπολογισμό, τάξεως ε, δισεκατομμυρίων βέβαια, αλλά θα έχει ε, επιγόντως επιπτώσεις και πολύ γρήγορα στις ε, ροές τις εμπορικές. Και ε, θα πρέπει επιγόντως να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Και τίθεται ένα κρίσιμο ερώτημα. Έχουμε προετοιμαστεί επαρκώς για ένα σκληρό Brexit χωρίς συμφωνία. Γιατί εμείς ανησυχούμε ειλικρινά. Και μπορεί να έχει πολλές συνέπειες για τις εμπορικές ροές και ο αγροτοδιατροφικός τομέας μπορεί να πληρώσει τα σπασμένα. Εσείς λοιπόν συμφωνείτε, συμμερίζεστε αυτή την ανησυχία μας και τι θα κάνετε. Γιατί ενδεχομένως να χρειαστούν μέτρα στήριξης για να αποζημιωθεί ο κλάδος. Και η Επιτροπή μας, Επιτροπή Γεωργίας το πρωί ψήφισε για ένα επιπλέον ε, προϋπολογισμό για υποστηρικτικά μέτρα. Ερωτώ λοιπόν μπορούμε να υπολογίζουμε και στη δική σας υποστήριξη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Υπουργό Λεπά που ήρθε σήμερα στη συνεδρίασή μας. Ε, έχουμε κοινέ ανησυχίες. Για παράδειγμα, το θέμα του προϋπολογισμού και την κατάσταση μετά το Brexit. Α, πάντως, διαρωτώ με μήπως αυτό που θα πρέπει να μας προβληματίσει κυρίως είναι τι είδους γεωργία θέλουμε στο μέλλον στην Ευρώπη, τι είδους τρόφιμα θέλουμε στο μέλλον. Και είμαστε έτοιμοι να ασχοληθούμε όλοι με το θέμα αυτό, γιατί για τις εμπορικές συμφωνίες, για παράδειγμα, αντιμετωπίζουμε τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα σαν να είναι τυχαία εμπορικά προϊόντα. Ενώ θα πρέπει να αρδεύουμε τις γεωργικές μας εκτάσεις για την οικονομία, για την ποιότητα των τροφίμων, για τον πολιτισμό μας, για τη γεωργία μας. Έχουμε κάποια μέτρα ώστε ε, από τα γεωργικά προϊόντα να διαχωρίζουμε κάποια και να τα χαρακτηρίζουμε γεωργικής ε, ε, στρατηγικής σημασίας και δεν είναι απλά εμπορικά προϊόντα, όλα τα γεωργικά προϊόντα. Ευχαριστώ κύριο Σρίστοφ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, ε, συμφωνώ με τις ανησυχίες κάποιων συναδέλφων. Σήμερα όλοι οι γεωργοί βρίσκονται σε διεθνή ανταγωνισμό. Εισάγουμε ανταγωνισμό λόγω των διεθνών συμφωνιών μας και οι δικοί μας οι γεωργοί είναι σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με εκείνους των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, επόμενη ΚΑΠΑ δεν ε, προβλέπει... Ε, προβλέπει το, 2000, ε, το 2027 εξίσωση των ενισχύσεων. Μετά από τόσα χρόνια μετά την ένταξη έχουμε ακόμα αυτό το πρόβλημα. Επίσης η πανόλης των χείρων. Έκανα πρόταση να διατεθούν περισσότερα κονδύλια για να αντιμετωπιστεί η νόσος και να αναπτυχθεί εμβόλιο. Ελπίζω ότι οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2020 να εξελιχθούν ομαλά και μπορώ επίσης να υπολογίζω στην υποστήριξή σας για την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ, η κυρία Κρόνενμπεργκ. Κύριε Λίντσε, κύριε Υπουργέ Ελέπε. Έχουμε μια έκθεση όπου αναφέρεται μια ρίση του Γκάντι ότι το πώς αντιμετωπίζουμε τα δάση αντικατοπτρίζει το πώς αντιμετωπίζουμε ο καθένας τον άλλον. Και αν δούμε ότι ο η Αμαζονία φλέγεται εδώ και μέρες και κάθε μέρα με δραματική απώλεια ε, βιοπικιλότητας με τεράστιες εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα και θα πρέπει να δούμε μετά την ολοκλήρωση της πυρκαγιάς τα προβλήματα που θα προκύψουν για να ε, απελευθερωθούν τεράστιες εκτάσεις για βιομηχανική γεωργία. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Τους επόμενους έξι μήνες θα πρέπει να περιμένουμε ε, μεγάλες αλλαγές και ε, ε, εμείς ήδη έχουμε ακούσει την Επιτροπή να κάνει νέες δηλώσεις. Πιστεύετε ότι με βάση τον αλληλοεξαρτώμενο και δικτυωμένο κόσμο δεν θα έπρεπε να ε, τροποποιήσουμε και την πολιτική μας ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες αλυσίδες που διαμορφώνονται στην γεωργική πολιτική και την πολιτική τροφίμων. Ε, ίσως στο Μερκοσούρ θα πρέπει να ε, δράσουμε βέβαια. Δεν έχουμε πολύ μεγάλη δυνατότητα επιρροής ε, για να επιβάλλουμε τις αρχές μας για τη βιωσιμότητα. Εσείς είπατε ότι θέλετε να απλοποιήσετε την ΚΑΠ. Ε, θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τη ε, διατήρηση της βιοπικιλότητας με την πολιτική για την καταπολέμηση του κλίματος και τη σωστή πολιτική τροφίμων που θα κάνουν τη διαφορά. Ευχαριστώ. Κύριε Κούσμιουκ. σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, υιοθέτησε ψήφισμα σημαντικό που περιλάμβανε και την προσδοκία τα κονδύλια της ΚΑΠ στο επόμενο ΠΔΠ να παραμείνουν αμή άλλο στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο ΠΔΠ 2014-2020. Ποια είναι η άποψη της Φιλανδικής Προεδρίας επ' αυτού. Και μια άλλη ερώτηση. Αναφέρθηκε αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι στην Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Μερκοσούρ. Για παράδειγμα, οι γεωργοί στι χώρε ε, Μερκοσούρ χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα που απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την ε, εισαγωγή τέτοιων προϊόντων ε, δεν θα δημιουργηθεί απειλή κυρίω για τους παραγωγού βοήου κρέατος και πουλερικών με προϊόντα που θα εισάγουμε και που θα έχουν παραχθεί με ουσίες που εδώ απαγορεύουμε. Επίσης, η ε, ε, κτηνοτρόφοι το χωρών κοσουρ δεν κόπτονται και ιδιαίτερως για την καλή μεταχείριση των ζώων. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ε, έχουμε καλύτερη εφαρμογή των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, γιατί αν τηρήσουν τις δικές μας προδιαγραφές θα γίνουν πιο υψηλές τιμές των προϊόντων τους και θα χάσουν ανταγωνιστικότητα. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό. Κύριε Αγγιλέρα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας προηγουμένως και στην Επιτροπή Αλίας. Ε, σήμερα είχα τρεις ε, επιτροπές και έτρεχα από τη μία στην άλλη. Δεν με διευκόλυνε το πρόγραμμα το σημερινό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, πρώτη μου ανησυχία για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε περικοπές στα κονδύλια της ΚΑΠ. Εσείς ως μέλος της φιλανδικής ε, κυβέρνησης Είστε υπέρ της διαφύλαξης του γεωργικού προϋπολογισμού ή και γενικώ για τη διαφύλαξη των ε, επιπέδων των κονδύλων του ΠΙΔΑΛΤΑΠΗ. Είναι σημαντικό να μάθουμε τη θέση της φιλανδικής κυβέρνησης. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε 1,3% του ακαθάριστου χώρου εισοδήματο των κρατών μελών για όλες τις πολιτικές και για να διαφυλάξουμε τα κονδύλια όλων των πολιτικών και όχι μόνο της ΚΑΠ. Επίσης, μεταβατικός κανονισμός, σημαντικός, όσο και να επισπεύσουμε την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ αποκλείεται να την υλοποιήσουμε πριν το 2023, για να μην, μέχρι το 2022, για να μην πω το 2023. Ο μεταβατικός κανονισμός είναι ήδη απαραίτητος από τώρα. Πιστεύετε ότι θα ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις αυτές. Επίσης, αναφερθήκατε στη μικροβιοική αντοχή. Έχουμε σημειώσει μεγάλη νομοθετική πρόοδο. Έχουμε δύο κανονισμούς ε, για τα, για τις, ε, ε, για τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις ζωοτροφές, τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Οπότε έχουμε ήδη σημειώσει πρόοδο, γιατί μερικέ φορέ δεν είναι αντίθετη εντύπωση. Τώρα για τι εμπορικέ συμφωνίε, είτε με τη Μερκοσούρ είτε με την Νότια Αφρική, δεν θα πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά την ευρωπαϊκή περα... παραγωγή. Κάτι που γίνεται, γιατί υπάρχει ανισότητα των προδιαγραφών. Ε, αυτό έχουμε στην Νότια Αφρική με τα σπεριδοειδή, στο Βιετνάμ με το ρύζι, ε, με, στο Μερκοσούρ με άλλες παραγωγές. Πώς θα εξασφαλίσουμε αυτή την ε, διόρθωση της αδικίας, γιατί οι Ισπανοί γεωργοί και οι Ευρωπαίοι γεωργοί γενικώ ε, θεωρούν ότι χάνουν δυσμενού μεταχείριση από τέτοιε εμπορικέ συμφωνίε. Συνάδελφε Αντέμου. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, Πολλές, ε, υπο, πολλές πυρκαγιές είναι ένα επίκαιρο θέματα και βέβαια δεν είναι θέμα τωρινό, είναι παλιό. Ε, θέμα παλιό και για τη χώρα μου τη Βουλγαρία και για πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είπατε ε, ότι τα προληπτικά μέτρα είναι πολύ σημαντικά εδώ. Η Φιλανδία τι μέτρα έλαβε, τι έχει λάβει σε αυτό το τομέα. Συνάδελφε Αμάρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, όλοι γνωρίζουμε ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που θα ισχύσει σε 28 χώρες μέλη με τόσο διαφορετικά γνωρίσματα είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Το είπατε κι εσείς, το είπαμε κι εμείς, ότι υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ της χρηματοδότησης της πολιτικής ε, και της ε, επιθυμίας μας να φέρουμε τους γεωργούς στο επίκεντρο της τροφικής αλυσίδας. Και έχουμε και την ε, κυριαρχία, την εθνική κυριαρχία. Όταν μιλούμε για ε, γεωργική παραγωγή, ουσιαστικά μιλούμε για κυριαρχία και αυτό θέλει να κάνει, επιστηστική κυριαρχία. Αυτό θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ καλά. Βέβαια αυτά τα θέματα είναι συναφή με, το, με τη χρηματοδότηση. Είναι αλληλένδετα μεταξύ του. Εγώ δυστυχώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με την αισιοδοξία σα. Δεν συμμερίζομαι την θετική σα αντίληψη. Και παρά το εντατικό έργο τη Επιτροπής, του Επιτρόπου, του Αρμόδιου για τη Γεωργία και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα στη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας. Μακάρι να γινόταν, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να εστερνιστώ την αισιοδοξία σας. Μπορείτε να με καθησυχάσετε ε, α, ότι αν υπάρξουν προτάσεις για περικοπή του γεωργικού προϋπολογισμού, ο Φιλανδός τουλάχιστον υπουργό θα αντιταχθεί σε μια τέτοια πρόθεση. Ευχαριστώ κύριο Σαβαρμά. <clears throat> Ευχαριστώ Νόρμπερτ. Καταρχήν ε, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη που άργησα να έρθω. Έπρεπε γιατί ήμουν ο υπεύθυνο για τη διαδικασία δημοσιονομικής απαλλαγής και αυτό πήρε χρόνο. Όμως θα κάνω μία εξαίρεση και σε 7,5 χρόνια θα μιλήσω φιλανδικά. Αγαπητέ Υπουργέ, είναι μεγάλη χαρά που σας βλέπουμε πάλι εδώ ε, συγγνώμη και πάλι που άργησα λόγω άλλων υποχρεώσεων. Η ερώτησή μου αφορά επίσης ε, τα χρήματα. Τα τελευταία πέντε χρόνια είχα την τιμή να είμαι ο πρώτος αντιπρόεδρος ε, της Επιτροπής του Προϋπολογισμού και είχα πολλές ευκαιρίες εκεί να συζητήσω με τον Επίτροπο Έτιγκερ επιθεμάτων που αφορούν τη γεωργία. Ε, τώρα πρέπει να δούμε την ευρύτερη εικόνα. Έχω την εντύπωση ότι αν δούμε τις προκλήσεις με τις εμπορικές πολιτικές, αν δούμε τις πολιτικές για το κλίμα, ή ε, τέλος πάντων την ευρύτερη εικόνα, αν κάνουμε τώρα περικοπές ε, είναι δύσκολη η επιλογή. Ρωτώ το εξή και συμφωνώ με τη συνάδελφα Αγγιλέρα εδώ. Η χώρα που ασκεί την Προεδρία ε, μπορεί να δώσει το παράδειγμα εδώ, γιατί νομίζω ότι είναι προς το κοινό μας συμφέρον να μην κάνουμε περικοπές στη γεωργία, έτσι όπως έχουν τα πράγματα παγκοσμίως. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρίστοτσεν. Χωρίς μικρόφωνο. Συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Ε, τρία αιτήματα από τους Δανούς ε, και από μένα. Να είστε απλοί, να είστε απλοί, να είστε απλοί. Μάλιστα. Ε, η πιο σύντομη παρέμβαση σήμερα το απόγευμα. Και τελευταίος παρεμβαίνων... Α, όχι. Ε, έχουμε και η πρώτη τελευταία, η κυρία Σάιντεχόφερ. Ναι, και εγώ είμαι υπέρ της διευκόλυνσης της ε, ε απλούστευσης. Νομίζω ότι η Φιλανδική Προεδρία θα ε, επιτελέσει πρόεδρο, ε, πρόοδο στον τριμερή διάλογο για την ΚΑΠ. Ε, συνεχώς μπαίνουν νέα στοιχεία, στρατηγικό ε, στρατηγικός σχεδιασμός για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, ορισμοί για την αποτελεσματική γεωργική παραγωγή. Αυτά βέβαια δεν είναι απλούστευση. φοβόμαστε μήπως γίνουν πιο σύνθετα τα πράγματα. Μπορείτε να φανταστείτε ένα πιο απλό ε, μέλλον που θα απλουστεύσει την ΚΑΠ. Επίσης, ε, δώσατε ενίσχυση στην Βραζιλία. Ο πρόεδρος Μπολσονάρου τι, πώς αντέδρασε, είπε ναι, όπως ελπίζομαι. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Τίτο. Ευχαριστώ πρόεδρε, ο κύριος Μπιτό. Ευχαριστώ Υπουργέ που ήρθατε να μας μιλήσετε εδώ είμαστε όλοι για να προσπαθήσουμε να χτίσουμε μια γεωργία που να μπορεί με αξιοπρέπεια να ανταμείβει τους γεωργούς και τους αγρότες και ταυτόχρονα να ε, ε, καλύπτουμε ανάγκες πιεστικές που είδαμε στις τελευταίες εκλογές για το κλίμα, τη βιοπικιλότητα, τη διαφύλαξη των γεών. Εμείς που είμαστε αγρότες όταν κατεβαίνουμε ε, από το τρακτέρ μας ε, θα πρέπει να μπορούμε να πιάνουμε τη γη, το χώμα και να είναι καλό αλλά και η γη ευρύτερα με γάμα κεφαλαίο ο πλανήτης μας ε, θα πρέπει να δούμε ότι η οικολογία δεν είναι αντιμέτωπη με την οικονομία ε, έχουμε την εντύπωση ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να συγκλίνουν. Αν δούμε όμως αντικειμενικά και από κοντά τα πράγματα θα διαπιστώσουμε ότι οι δομές που μιλούν για την αγροοικολογία είναι δομές ε, ε, ε, άκρος ανταγωνιστικές που επιτρέπουν στους αγρότες να έχουν περισσότερο εισόδημα σε μια λογική παραμένοντας όμως σεβασμού και ισορροπίας για τους πόρους και εδώ σκέφτομαι το νερό που θα κυριαρχήσει στο μέλλον που σέβονται τη βιοπικιλότητα, το κλίμα και την υγεία των καταναλωτών. Α το σκεφτούμε λοιπόν, ας οικοδομήσουμε εκείνε τι δημόσιε πολιτικέ που υποστηρίζουν ειδικά αυτή την ανάπτυξη και κυρίω. Έγινε λόγο για τη γεωργία, για την απασχόληση και για την εγκατάσταση των νέων. Κοιτάξτε πώς δίνετε τις ενισχύσεις της ΚΑΠ ε, που είναι στρεματική ενίσχυση. Δηλαδή όσο περισσότερα στρέμματα έχεις, τόσο περισσότερη ενίσχυση και όσο πιο πολλά λεφτά παίρνεις, αγοράζεις και άλλα στρέμματα ή εκτάρια. Έτσι έχουν χαθεί στη Γαλλία σε 20 χρόνια μισή αγρότες. Μήπως να γίνει διαφορετικά η δημόσια στήριξη της κοινή γεωργικής πολιτικής και όχι με βάση την επιφάνεια, αλλά με βάση τις θέσεις απασχόλησης, με τη μονάδα απασχολούμενου. Γιατί έτσι θα απελευθερωθεί και η γη, γιατί δεν θα είναι το κίνητρο να αγοράζει γη για να παίρνει λεφτά, αλλά η απασχόληση. Και το απλουστεύω λέγοντας ότι αυτό θα μπορούσε να είναι και ένας τρόπος απλούστευσης που ζητάνε πολλοί συνάδελφοι εδώ τη κοινή γεωργικής πολιτικής. Και ένα τελευταίο για το Brexit. Εδώ ανησυχούμε όλοι για τις επιπτώσεις του Brexit. Σήμερα το πρωί ψηφίσαμε μέτρα για μια-δυο χώρε και θα παρακαλούσα ή δυνατόν να έχουμε γενική συνολική προσέγγιση γιατί δεν θα επηρεάσει μόνο την Ιρλανδία, τη χώρα του κυρίου Χόγκαν δηλαδή, το Brexit. Ευχαριστώ. Είστε τυχερός, έχουμε λίγο χρόνο. Ε, θα είμαι πιο αυστηρός ε, αργότερα στην τήρηση του χρόνου. Ο κύριος ε, Γιάρ, τελευταίος, ευχαριστώ πρόεδρε, υπουργέ, συμπληρώνοντας τους συναδέλφους δύο ερωτήσεις και μία παράκληση. Ερώτηση πρώτη για την έρευνα, για την κοινωνική, τεχνολογική πρόοδο, ίντερνετ, νέες μέθοδοι εκτροφής, ε, αυτόνομες μηχανές. Αυτό θα το φροντίσετε στη Γεωργία γιατί δεν θέλουμε νέους αγρότες, γιατί πιστεύουν περισσότερο ότι αυτά είναι παλιά οικονομία, όχι καινούρια, όχι. Χρειαζόμαστε και έρευνα και τεχνολογία. Δεύτερη ερώτηση, άμεσες πληρωμέ. και πώς αυτές διαμορφώνεται. Τονίζεται συνέχεια με ΑΙ ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και εμείς φροντίσαμε αυτές να μειωθούν στην Επιτροπή μας. Πλην όμως αναγκάστηκα να διαπιστώσω ότι υπάρχουν διαφορές και μεταξύ των περιφερειών στα ίδια τα κράτη-μέλη και αυτές είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι μεταξύ των κρατών μελών. Ε, θα ασχοληθείτε και με την ε, δικαιοσύνη. Γιατί έχουμε χώρες όπου στο Νότο είναι 200 ευρώ το εκτάριο ενίσχυση 500 και στο Βορρά 50. Και το τρίτο, η παράκληση. Ε, καθυστέρησα λίγο γιατί ήμουν στην Επιτροπή Αναφορών όπου ε, αποφασίσαμε να γίνει ακρόαση για το λύκο. Ε, ποιο είναι ο πληθυσμό των λύκων. Το Δεκέμβριο θα γίνει ακρόαση, ενδεχομένω μαζί με την δική μα Επιτροπή εδώ και την Επιτροπή Περιβάλλοντο. Αν έχετε κανέναν καλό εμπειρογνώμονα εγνωσμένου κύρου και κοινή αποδοχή, θα σα ήμουν ευγνώμων. Γιατί θα είναι και παραμονές των Χριστουγέννων και θα έχει γνωρίσει έτσι, μεγάλη δημοσιότητα η ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ. Δύο μιλητέ υπάρχουν ακόμα. Συνάδελφε Τσόιντερ και Άφραμ και κανέναν άλλον. Κλείνω λοιπόν εδώ τον κατάλογο των ομιλητών. Στις 5 πρέπει να φύγει ο υπουργό και πρέπει να προλάβει και να απαντήσει. Όχι. Α, η συνάδελφος Άφραμ. Ε, ε, συγγνώμη, Υπουργέ Λέπε, εδώ είμαι. Νομίζω ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τη μετάφραση. Ρώτησα για τα 10 δις και την έρευνα, αλλά όχι ε, πώς θα τα δαπανίσετε. Ε, αναφέρθηκα στις διαφορές μεταξύ χωρών και αν μπορούμε να βρούμε μια ε, λύση ώστε οι χώρες που έχουν καλύτερη έρευνα να μοιράζονται τα δεδομένα τους τα ερευνητικά με τις χώρες που έχουν χαμηλότερο επίπεδο έρευνας. Αυτό, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ε, πάμε στην τελική απάντηση μετά τον τελευταίο γύρο ερωτήσεων από τον Υπουργό. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Ας αρχίσουμε με τους νέους αγρότες και πώς βλέπω εγώ το θέμα. Νομίζω ότι για τρίτη φορά το λέω. Οι νέοι ε, αγρότες, ε, είναι νέοι γεωργοί, είναι πολύ σημαντικοί για μας. Είναι σημαντικό να έχουμε νέους γεωργούς στην Ευρώπη. Και γι' αυτό υπάρχουν και μέτρα στήριξης ε, που πρέπει να συνεχιστούν στη νέα ΚΑΠ. Επίσης, πρέπει να προβλέψουμε υποστήριξη για τις επενδύσεις, μορφές ευέλικτες, ε, επίσης η διαδοχή είναι πολύ σημαντική στις εκμεταλλεύσεις και η εκπαίδευση, η κατάρτιση των γεωργών είναι πολύ σημαντικό θέμα. Οι νέοι γεωργοί χρειάζονται νέες δεξιότητες ε, για να βελτιώσουν την παραγωγή. Προφανώς η παραγωγή πρέπει να είναι κερδοφόρος και χρειάζεται κερδοφόρος γεωργία. Γι' αυτό θα ε, προσελκυστούν ε, στη γεωργία. Αυτό είναι ένα κίνητρο, αλλά χρειάζονται και στοχευμένα μέτρα. Τώρα για τα μεγάλα αρπακτικά ζώα Τώρα έχουμε γίνει δικοί στους ε, λύκους. Για τους λύκους ρωτήστε μας ό,τι θέλετε. Πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση αυτή. Ε, είναι σαφές. Και η σημερινή συζήτηση είναι ένα κομμάτι του τι πρέπει να γίνει. Τώρα για το Brexit ε, θα κάνω μερικές παρατηρήσεις εδώ. Στην περίπτωση του Brexit είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε με μια ε, νέα βρετανική κυβέρνηση για να αποφύγουμε το σενάριο της μη συμφωνίας, να έχουμε όσο γίνεται πιο στενές σχέσεις στο μέλλον, ε, όσο πιο πολύ γίνεται. Είχαμε ε, πικρές εμπειρίες από διαταραχές, αναταράξεις στην αγορά στο παρελθόν και θα τις αποφύγω με πασή Καταλαβαίνουμε απόλυτα τις ανησυχίες σας σε σχέση με τις αναταράξεις στην αγορά, ε, στις αγορές εν ώψη του Brexit. Αυτό το αντιμετωπίζουμε και αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά τις ανησυχίες σας. Δεν παρακολουθούμε μόνο το, τις επιπτώσεις ε, στο, του, του Brexit βέβαια και η Κομισιόν προφανώς θα αναλάβει τις απαραίτητες δράσεις. Η Κομισιόν έχει μια διευρυμένη εντολή να προβεί στη, στα κατάλληλα μέτρα ε, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία. Και Είμαι βέβαιος ότι η Κομισιόν θα αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες και δυνατότητες που έχει. Αυτό είναι σαφές. Προφανώς και συμφωνώ πάρα πολύ στην προτεραιότητα της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Ε, Εμεί έχουμε υψηλό επίπεδο εδώ, υψηλά πρότυπα και Ε, για να μην παρεξηγηθώ, επαναλαμβάνω αυτό που είπα, ε, το μοίρασμα, ο επιμερισμό των ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Τώρα, για την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων, αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ σοβαρό πρόβλημα και ε, συμφωνώ με τις αποφάσεις σας πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη. Γιατί έχουμε δει πόσο περισσότερο στοιχίζει η αντιμετώπιση των κρουσμάτων. Ε, χρειάζονται ε, πολλές διασφαλίσεις για να ε, περιορίσουμε τη μόλυνση καλύτερες συνθήκες υγιεινής, ε, στις μεταφορές. Ε, ε, εδώ όλα είναι σημαντικά. Τώρα για το, τις πυρκαγιές στην Αμαζονία, πολύ, τεράστιο θέμα όπως και γενικότερα η αποψήλωση των δασών. Έχουμε εδώ μια έκθεση της Κομισιόν από τον Ιούλιο, που είναι μια καλή βάση για να στηρίξουμε τη βιώσιμη χρήση της γης, βιώσιμη δασοπονία, ανανέωση των δασών, ε, καταπολέμηση της αποψήλωσης των δασών. Ε, τις νόσους ε, των ε, δασών, των δέντρων και των φυτών. Αυτά όλα είναι παγκόσμια προβλήματα. Σε όσο καλύτερη κατάσταση είναι τα δάση, τόσο περισσότερο θα παίζουν τον ρόλο τους. Στη Φιλανδία, εδώ και δεκαετίες, η δασική πολιτική στηρίζεται στην αρχή ότι θα πρέπει να ε, έχουμε μια οικονομική εκμετάλλευση του δάσους που θα μας επιτρέψει να το γνωρίσουμε, θα μας επιτρέψει να το προστατεύσουμε με ε, αντιπυρικές ζώνες. Έχουμε βεβαίως και ε, πτήσεις παρακολούθησης της κατάστασης στα δάση. Αυτά είναι τα μέτρα που έχω υπόψη μου. Η... Ναι, προσφέρθηκε βοήθεια στη Βραζιλία, αλλά δεν είμαι βέβαιος για την απάντηση. Ε, πράγμα που δείχνει ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να αξιοποιεί τα διαθέσιμα εργαλεία για την πρόληψη. Και το ίδιο ισχύει και για τις εμπορικές συμφωνίες. Ε, το είπα και το ξαναλέω. Δεν μπορούμε να έχουμε συμφωνίες με κάθε τίμημα. Υπάρχει ένα σημείο καμπής. Θα πρέπει να αναδείξουμε τα κρίσιμα ζητήματα πριν προχωρήσουμε σε εμπορική συμφωνία και να τα εκφράσουμε. Να μην υπάρχουν αναταράξει στην αγορά, να μην ε, υποβαθμίζεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, να μην ε, ε, μειώνεται. Δεν μπορούμε λοιπόν με κάθε τίμημα να προχωρούμε σε εμπορικές συμφωνίες. Γνωρίζω πολύ καλά ε, αυτό που είπατε για τα εντομοκτώνα και τα ζυζανιοκτώνα ε, που διαφέρει η χρήση τους εκεί από ό,τι εδώ. Επίσης η μικροβιακή αντοχή είναι διαφορετική εκεί από ό,τι εδώ. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας πριν προχωρήσουμε σε σύναψη συμφωνίας. Υπάρχουν ε, κάποια κρίση. Αυτά είναι τα κρίσιμα σημεία. Τώρα για τη χρηματοδότηση και τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Το σημαντικό είναι να έχουμε μια δημοσιονομική πρόταση ισορροπημένη που θα προάγει την ΚΑΠ και να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των ε, αναγκών και των μηχανισμών στήριξης. Δεν μπορεί δηλαδή να αυξάνονται οι απαιτήσει και να μειώνεται η χρηματοδότηση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό το λέω εξ ονόματος της Φιλανδικής Προεδρίας. Επίσης, ε, το έχω πει πολλές φορές. Έλαβα ε, ηχηρό το μήνυμα από εσά σχετικά με τη μη μείωση της χρηματοδότησης και θα ε, ε ενημερώσω τον Φιλανδό Πρωθυπουργό. Το θέμα ε, είναι δικό μου έμεσα μόνο, είναι θέμα άμεσα του Πρωθυπουργού και σας υπόσχομαι ότι θα λάβει ηχηρό ε, το μήνυμα που στέλνετε. Τώρα, η απλούστευση είναι απόλυτα αναγκαία και έχουμε δεσμευτεί υπέρ της πραγματικής ε, απλοποίησης. Είμαστε ε, υπεύθυνοι όλοι εδώ, σε κάθε χώρα, κάθε Υπουργείο. σε κάθε μεταρρύθμιση. Μπορούμε να λάβουμε καλύτερα υπόψη τις διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Κάποιος με ρώτησε ε, για τη διαφοροποίηση της πολιτικής μέσα στο ίδιο κράτος μέλος. Η ΚΑΠ περιλαμβάνει και τις δύο διαστάσεις και είναι καλό που έχουμε προτάσεις που επιτρέπουν τη, και τους δύο τύπους ισορροπίας και ε, ευθυγράμμισης των κρατών μελών. Επίσης, η σημασία του καθαρού αέρα, καθαρού νερού. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση για καλά τρόφιμα, βιωσιμότητα, ανάπτυξη των δασών. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ για την τροφή για σκέψη που μου δώσατε. Ε, τα κατέγραψα αυτά που μου είπατε και θα ε, προωθήσω στους συναδέλφους μου όλη αυτή την ενημέρωση. Επίσης, ε, οι προϊστάμενοι μου θα ενημερωθούν σε σχέση με τα αιτήματά σας για την χρηματοδότηση και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε μια καλή κοινή γεωργική αγροτική πολιτική και να βρεθούν επικοδομητικές λύσεις ε, που θα εξασφαλίζουν το μέλλον ε, διατηρώντας ε, απασχόληση και είναι σημαντικό βεβαίως εδώ να διατηρήσουμε τους νέους γεωργούς. Ευχαριστώ. Frau Kollegin Aguilera, bitte.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 Ε, το, το μέλλον της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Ε, όλοι προσβλέπουμε στην καλύτερη δυνατή λύση και η συνάντηση αυτή έδειξε μετά τη συνάντηση του Ιουλίου για τις εμπορικές συμφωνίες ότι αυτό το θέμα απασχολεί πολλούς συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ ε, αισιόδοξο για μια καλή συνεργασία τους επόμενους μήνες. Καλή, ότι θα έχουμε ε, ε, καλή επαφή μέχρι το Δεκέμβριο για να προχωρήσουν όλα τα θέματα που αναφέραμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.